Καλησπέρα συναδελφοί, άρχεται εκ νέου η συνεδρίαση. Να σας ενημερώσω καταρχάς ότι τα πρακτικά της χθεσινής ε, συνεδρίασης είναι διαθέσιμα. Αν έχετε σχόλια. Αλλιώς εγκρίνονται. Ξεκινούμε την απογευματινή μας